Hello everyone. Good evening. Καλησπέρα σα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. This evening, even though we are, we know... Καθίστε. Ξέρουμε ότι έχουμε έρθει να ψηφίσουμε όμως. Επειδή εξακολουθεί να είναι συνεδρία τη Επιτροπής, πρέπει πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, αν κάποιος ε, δεν διαφωνεί, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Να σας πω επίσης ότι έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος για την αλλαγή χρήσης γης στο LULUCF στις 19 Οκτωβρίου και έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα πιο σημαντικά πολιτικά ζητήματα που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Η συζήτησή μας ε, βασίστηκε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου και βεβαίως ε, έχουμε και τη γενική προσέγγιση της 16 Οκτωβρίου του Συμβουλίου. Η πρώτη συνεδρίαση περιορίστηκε απλώ στην παρουσίαση των αντίστοιχων θέσεων και δεν ελήφθη κάποια απόφαση επί του περιεχομένου. Αποφασίστηκε τα περισσότερα θέματα να τα εκχωρήσουμε σε τεχνικό επίπεδο για περαιτέρω συζητήσεις πριν γίνει ο δεύτερος τριμερής διάλογος. Θα σας ενημερώνουμε γι' αυτά και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε στο προκείμενο για απόψε. Ψηφοφορία για την πρόταση οδηγίας για την πρόθεση της χρήσης ε, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πρόκειται για αναδιατύπωση και ο εισηγητής είναι ο κύριος Άικχαουτ και πραγματικά θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ησυχία γιατί τα πράγματα είναι περίπλοκα. Όχι εσείς κυρία Άικχοτ, εσείς έχετε την έκθεση, εσείς μπορείτε να μιλήσετε. Στους υπολείπους απευθύνομαι. Οι σοσιαλιστές είναι λαλίστατοι σήμερα. Ανησυχείτε. Εντάξει, να το σκέφτεστε σιωπηλά. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε λοιπόν συμβαστική τροπολογία περιθμών 1. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να γίνει μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Σας παρακαλώ λίγη υπομονή μέχρι να βρούμε και το τεχνικό. Συγγνώμη, πρέπει να περιμένουμε γιατί το μηχάνημα δείχνει εντελώ άλλα αποτελέσματα. Δείχνει ότι είναι η φιλελεύθερη εδώ, είναι η ομάδα των φιλελευθέρων αυτή που συνεδριάζει εδώ στην αίθουσα και δείχνει σαν να είστε όλοι φιλελεύθεροι εδώ. Νομίζω ότι λέει ότι έχει 18 σοσιαλιστές επιπλέον. So ε, πέρας και ξαναψηφίσουμε. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. out my hands, so we have to wait a Συγγνώμη, πρέπει να περιμένουμε να πάει ο τεχνικός ε, στην καμπίνα. Έτσι το είπε, καμπίνα. Για να αλλάξει και αντί για αίθουσα των φιλελευθέρων να είναι αίθουσα της Επιτροπής Περιβάλλοντος εδώ. Συγγνώμη, δεν φταίω εγώ, ξέρω ότι βιάζεστε. It's okay. Can you it's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 Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να ξαναδοκιμάσουμε. Συγγνώμη. Ήρθα τρεχάλα και ξέχασα την, ολομέλεια, την κάρτα μου στην Ολομέλεια. Θα ψηφίζω με ανάταση χειρός. Έχω στείλει τον βοηθό μου. Ναι, ναι. Έχω στείλει κάποιον να τη φέρει. Έχουμε δύο περιπτώσεις, επομένως θα πρέπει να ψηφίζουμε και θα μετράμε δύο ψήφους με ανάταση χειρός. Απλώς να μας δείχνετε λοιπόν αν ε, είστε υπέρ κατά. Uh, Συμβαστική τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Από το ECR έχουμε έναν περιττό το ECR πρέπει να αφαιρέσει μία κάρτα. Εντάξει είμαστε τώρα, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3α. 3A. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σελίδα 6, τροπολογία 391. Ποιος είναι υπέρ. Κατά της 391. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πίτερ, μπορείτε να μας δείξετε τι ψηφίζετε. Ωραία, ευχαριστώ. Πέρασε τη ψηφοφορια Εγκρίνεται. 394 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 397 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 398 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 400 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 402 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 403 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 404 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 405 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 405. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία ψηφοφορίας εγκρίνεται. 406 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση γιατί 408 άρχεται η ψηφοφορία. Ένας της πληροφορίας εγκρίνεται 33-32. 410 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 411. Καταπίπτει. 412. Ποιος είναι υπέρ της 412. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 413. Συγγνώμη, 414. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 416 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 415 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 420 και 421 μαζί υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για τις 420 και 421 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 422 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 423 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 424 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 425 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 426 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 427 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε προς τη σελίδα 15 για τη συμβαστική τροπολογία 4α. Υπέρ της 4α. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 4α. Άρχεται ψηφοφορία. And it is uh, closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Compromise b Συμβαστική τροπολογία 4β. Who is in favor? Υπέρ. Ή μάλλον πάμε ηλεκτρονικά. Επειδή είναι συμβαστική τροπολογία, καλύτερα να κάνουμε την επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Come to the amendments. Πάμε στις τροπολογίες. Συμβαστική τροπολογία 6 πρώτα. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εδώ έχουμε ένα block A το οποίο ξεκινάει με την 465 υπέρ του block A κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 464. Έχουμε τέσσερι τροπολογίε, την 464, 466, 475, 476. Ποιο είναι υπέρ αυτών των τεσσάρων. Κατά, αποχές απορρίπτονται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 467 υπέρ. Υπέρ της 467 κατά. Αποχές απορρίπτεται. 468 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 469 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 470 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 471 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 472 υπέρ όχι καταπίπτει Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μισό λεπτό να δούμε τι καταπίπτει, τι παραμένει. 4,81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4,77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 477. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 482 υπέρ 482 κατά αποχές απορρίπτεται 483 υπέρ κατά επαλήθευση για την 483 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 485 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 486 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 487 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 488 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 489 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 4.90 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρασε εγκρίνεται 4.91 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4,92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4,93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Δεν είδα καθόλου το άλδε. Που είναι σχετικό για την ισορροπία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 4.94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.95 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 496 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 497 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 498 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 499 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 499. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 500 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 501 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5... Αλλά να ελέγξουμε. Την 501. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 502 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 503 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 504 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 505 και 33 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 34 καταπίπτει. 506 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 508 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 509 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 510 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 511 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 512 υπέρ όχι καταπίπτει 35 και 513 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 514 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 515 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 516 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 517 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 517. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 518 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 519 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία στην 520, στο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 521 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μαζί με την 522 αυτό 523 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 524 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 525 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 526 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 527 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 528 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 529 υπέρ. Κατά. Αποχές απο... εγκρίνεται. 530 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 531 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 532 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 533 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 536 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 534 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.34. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 5.35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 539 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 540 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 541 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 543 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 542 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 5.44 και 45 και 46 είναι όμοιας υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Don't go too far. Μην πάτε μακριά. 558. 558. Σελίδα 27. Εδώ αυτό βλέπω. 558. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 551 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 552 υπέρ και 554 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 559 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 560 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 561 υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. 564 maybe? ...565 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 566 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 560 7 και 3.15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έχουμε κάποιες πανομοιότυπες, 5,78, 1000 κάτι, είναι unblock, όλα μαζί. Ποιος είναι υπέρ αυτού του block. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Την τροπολογία 578 και όλες τις υπόλοιπες που είναι μαζί της. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίες απορρίπτεται. 38 και 83 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5,71 υπέρ. Κατά. Α, δεν ήταν ξεκάθαρο. Ξανά. 5.71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Δεν καταλαβαίνω. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Περνάμε μια σελίδα. 580. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 581. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 579. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 583. Υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 584 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 585 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 588 και 589 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 591 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 592 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 590 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 587 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 594 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 594. Άρχεται η ψηφοφορία. Και κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 596-93 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 597 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 601 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 602 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 603 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 604 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 598 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 599 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 600 υπέρ Α, όχι, καταπίπτει. Είδα, όχι, είναι πανομοιότυπη. Η 41 καταπίπτει. 614 υπέρ κατά αποχές δεν είδα το ΕΛΚ 614 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 615 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 617 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 619 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 620 υπέρ. Μα είναι πανομοιότυπη. Συγγνώμη. Ήταν σε άλλη σελίδα και δεν το είδα. Η 621. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 622 υπέρ. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 616 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 622 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 624 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 625 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 626 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 627 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 628 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 629 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Όχι. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 631 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 632 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 632 άρχεται η ψηφοφορία. πέρα τη ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Πού είμαστε? 6.33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 και 639 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6.38. Όχι. Η 6.39 εγκρίθηκε. Προχωράμε λίγο. 6.40 υπέρ. Καταπίπτει. Then what? 6.41. Και ποια ακολουθεί τώρα 6.41. 641 και 642 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 648 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 643 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 644 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6.40 Πάμε στην 6.49 επειδή εγκρίθηκε η 6.44 υπέρ της 6.49 κατά ποχές απορρίπτεται. 6.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 651 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 653 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 654 υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται. 655 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 656 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 657 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48, 49 και 50 μαζί υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται εγκρίνονται αυτό μας οδηγεί πιο κάτω στην 665. 665 μαζί με 666 και 667 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τον μπλοκ αυτό. Ξέρω ότι είστε κουρασμένοι αλλά πρέπει να σηκώσετε τα χέρια σας για να είναι σωστή η ψηφοφορία. Άρχεται, πέρας. Εγκρίνονται, αλλά δεν σηκώσατε χέρια. Ωραία. Όταν εγκρίνεται πράγματα πάμε πιο γρήγορα. Ε, τώρα πηδάμε στην 677. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 677. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 679 ε, και 680 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 681 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5α υπέρ ποιος είναι υπέρ της 5α κατά αποχές να ελέγξουμε την συμβαστική 5α άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Αλήθεια λέει πρόεδρος 5β Υπέρ Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Απευθείας την 5β Άρχεται η ψηφοφορία για την 5β Παρακαλώ ψηφίστε. Δεν έχετε ψηφίσει όλοι. 5β. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πόπο. Ευχαριστεί η πρόεδρος. Σελίδα 62 περίπου, συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, υπέρ της συμβιβαστικής 7. Ευχαριστώ πολύ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Ας ε, ελέγξουμε, ας επελθεύσουμε. Στη συμβεστική 8 θέλουμε να δούμε αριθμούς, οπότε ψηφίστε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 980. 980 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 981 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2β Apparently it falls. Όπως φαίνεται καταπίπτει. Ωραία, πάμε στη συμβαστική 2α. 2α. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε παρακάτω, παραλείποντας πολλές τροπολογίες. Στη σελίδα 73. Η 984, ποιος είναι υπέρ. 984 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 985-986 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 987 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 988 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη 989 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 990 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 991 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 992 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 992 άρχεται ψηφοφορία It is closed. It is adopted. 993, 94, 95. Εγκρίνεται 9, 93, 94, Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 996 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 997 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 998 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 999 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Χιλιά δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Χιλιά τρία υπέρ κατά αποχές ας ψηφίσουμε με ανατασίχυρος 1003 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1004 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1005 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1006 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1007 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1008 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1009 υπέρ κατά 1009 παρακαλώ ποιος είναι υπέρ 1009 κατά εποχές απορρίπτεται 1010 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1011 μέχρι 1013 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1014 1014 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1015 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1016 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1019 υπέρ μαζί με τη 1020 κατά απορρίπτεται 1021 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1022 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί 1023 με 1026 ταυτόσιμες 1023 έως 1026 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 1027 κατά πέπτη 1027 ξεχωριστή ψηφοφορία για την πρόταση της Κομισιόν Έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία για πρόταση της Επιτρόπης σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 1028 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1000 να ελέγξουμε τη 1028 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ζήτω συγγνώμη 1029-1030 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 1031 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπλοκ, 1032 έως 1035 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 1041 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1042 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1045 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε τη 1045 ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1046 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1049 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1053 και 1064 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 1054 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 1054 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Η 10-21 εγκρίθηκε ή όχι. Πάμε στην 1058 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 1059 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1060 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1061 και 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 1062 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1065 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1066 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ομπλοκ 1067 έως 1070 Πέρα, κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τον μπλοκ αυτό ναι άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 1072 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1073 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πρέπει να ψηφίσουμε στις επόμενες 1104 ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1097 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Just a second to see. Ζητά ένα δευτερόλεπτο η πρόεδρος για να ελέγξει. let's vote on it and we can delete it <laughs> afterwards. It was rejected. 1098. 1098 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1099 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.02 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.03 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.08 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.09 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11.11 11, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται τέσσερα 120 και 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 120 να ελέγξουμε την 125, όχι. 127 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτω, ε, εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 όχι ναι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχή πίπτη μάλιστα έχετε δίκιο ναι, ε, εξαιτίας 151 ωραία καλά ναι αυτά πάμε στα 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 και 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ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 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ να ελέγξουμε την 191 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την 191. πέρας απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκατόν υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 206 υπέρ. Μισό λεπτό, πρέπει να το επαληθέσουμε αυτό, να δούμε αν πρέπει να ψηφίσουμε τη 12. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 200. Υπέρ της 200 κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208, 9 και 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε παλήθευση για τη 13. Ας την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. It's closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...219 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 220 υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 222 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 234 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ, κατά, 258. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν την είναι αυτή. 247 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκκρίνεται. 258 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για τη 258. The vote is open and... Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εκρίνεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ...279 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Και τελειώσαμε. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος θέλει το λόγο? Ο κύριος Γκερμπράντι κάτι θέλει να πει, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, πριν ε, ψηφίσουμε, μπορείτε να μας δώσετε λίγο χρόνο, κάποια λεπτά. Δύο-τρία λεπτά αρκούν. Θέλετε να διαβουλευτείτε. Εντάξει, δύο λεπτά. Να ρωτήσω τους υπολείπους αν σας επιτρέπουν δύο λεπτά. Δύο λεπτά σας παρακαλώ μη φύγετε, πρέπει να κάνουμε την τελική ψηφοφορία. Πέρασαν τα δύο λεπτά. Παρακαλώ καθίστε, αν θέλετε. Have the final vote. Για να γίνει τελική ψηφοφορία για την έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους. That concludes our meeting. Με αυτό ολοκληρώνεται η απόψινή συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε αύριο. Αλλά στην Ολομέλεια, όχι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ.